ιδίως στην Αστάνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει και θα υπομειστεί τις ευθύνες της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, λίγη εδώ αυτή η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο. Τώρα το επόμενο θέμα. Η έκθεση του Αγκουστίν Δίας Δεμέρα για τις τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι χρειάζονται βίζα θεώρηση. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο Μάλστρομ εδώ. Πολύ ευγενές το ότι προσήλθε την καθυστερημένη αυτή ώρα και θα δώσω αμέσω το λόγο στον εισηγητή μας, κύριο Κονσουέγκρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Θέλω να χαιρετήσω και την ομάδα εργασίας σας, αγαπητοί συνάδελφοι και συμπέθεροι. Ο κανονισμό 5039 κάθος 2001 καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χώρων υπό και των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων τη Ένωση καθώς και τον κατάλογο των χωρών, των άλλων χωρών, των οποίων οι πήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού 539 2001 που μας απασχολεί σήμερα έχει ένα τριπλό στόχο. Να μπορέσουμε να ενσωματίσουμε την Ταϊβάν στον θετικό κατάλογο, άλλες τρίτες χώρες και εδάφη όπως το Τρίτα και τον Πάκο Ανταλουσία, Σαν Λουθίνα, Γρεναδίσα, Δομίνικα, Γρανά, νησιά, Μάρσελ, Νικο, Μικρονησία και Παλάου να, ε, μετα, να τροποποιηθούν στον κατάλογο και επίσης να αντιμετωπιστεί το θέμα των νήσων Μαριάνας. Οι νήσοι Μαριάνας δεν παρουσιάζουν πρόβλημα γιατί οι κάτοικοί τους είναι Αμερικάνοι πολίτες. Σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες στις οποίες ανέφερα, η Κομισιόν δεν βλέπει λόγους για να αναστείλει την ανάγκη χορήγησης προξενική θεώρηση, βίζα, δηλαδή, ούτε και εμείς. Στην περίπτωση της Ταϊβάν έχει περάσει μια δημοκρατική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, μια ανάπτυξη στον οικονομικό, κοινωνικό και οικονομικό χώρο που είναι αξιέπαινη. Έχουν επιτέλους εδρεωθεί από το 1996 τα δημοκρατικά όργανα ξεκίνησαν οι πρώτες άμεσες δημοκρατικές προεδρικές εκλογές. Ο πρόεδρος, ο οποίος ε, εκλέγεται από όλους τους Ταϊφανέζους με καθολική ψηφοφορία, έχει θητεία τεσσάρων ετών και το Ζιάν που είναι η Βουλή της Ταϊβάν έχει 113 νομοθέτες. Από οικονομική άποψη η Ταϊβάν έχει μία, ένα από τα υψηλότερα κατακεφαλήν εισοδήματα στον κόσμο, 33.000 δολάρια. Η ανεργία ήταν μονάχα 5,2%, πολύ λιγότερη από το μεσόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεπερνάει το 10%. Το πρώτο τρίμηνο του 2010 η οικονομική ανάπτυξη ήταν 13,27 και το εμπορικό της ισοζύγιο ξεπέρασε το πλεόνασμα του ισοζυγίου ξεπέρασε τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτών. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2009, η Ταϊβάν είχε από οικονομική έποψη την 25η θέση στον κόσμο με ένα ε, ΑΕΠ 375 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρέπει να υπενθυμίσω το 2050 250 ήταν πιο φτωχή από την Ουγγάντα και από τη Δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, γιατί εξαρτιόταν μέχρι το 1960 από βασικά προϊόντα και εξαγωγές και βρισκόταν στην ίδια θέση με χώρες όπως η Κένια, η Νότια Αφρική και ο Λίβανο. Σήμερα όμως τα μεταποιημένα προϊόντα τη Ταϊβάν είναι πάνω από 97% των εξαγωγών της χώρας αυτής. Όπως είπα και προηγουμένω, με τον τρόπο αυτό έχει δημιουργηθεί και ένα ε, ρυθμός ε, που είναι μόνο 0,15%. Επομένως είναι σχεδόν μηδενικός ο αριθμός μεταναστών νομίμων ή παράνομων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι μόνο 40 περί παράνομοι μετανάστες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση προερχόντουσαν από την Ταϊβάν. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων, τα ηλεκτρονικά διαβατήρια της Ταϊβάν, πληρώνουν όλα τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, ICAO και η κατάσταση των Ταϊβανέζων στη διασπορά πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν διαβατήριο από τις αρχές της Ταϊβάν και είναι λογικό εφόσον χρειάζονται ειδικά κριτήρια για να έλθει κάποιος από το εξωτερικό στη Ταϊβάν, είναι λογικό να διατηρηθούν και αντίστοιχα κριτήρια για τους προερχόμενου από την Ταϊβάν. Για τα περισσότερα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτό από τη Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, δεν ζητά βίζα. Αλλά οι αρχέ τη Ταϊβάν έχουν δεσμευτεί να δώσουν πλήρη απαλλαγή για τι χώρε αυτέ από τι 11 Νοεμβρίου 2010, δηλαδή από αύριο, από σήμερα ουσιαστικά σχεδόν, σε ώρα Ταϊβάν. Αυτή λοιπόν η δέσμευση θα πρέπει να υλοποιηθεί όπω έχει ζητήσει και το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο, όμω επίση και οι μόνιμε αντιπροσωπείε των εμπλεκομένων τριών χωρών. Για όλους αυτούς τους λόγους κύριε Πρόεδρε και για άλλους λόγους που αναφέρω στη δεύτερη παρέμβασή μου πρέπει να δώσουμε αυτή την απαλλαγή από την προξενική θεώρηση στην Ταϊβάν όπως έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία. Σας ευχαριστώ τα μάλλα Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόβατσεφ για ένα λεπτό της Ευχαριστώ πρόεδρε, καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε Μάλστρομ. Η έκθεση του κυρίου Δίας Δεμέρα δείχνει ότι μετά από ολόκληρες δεκαετίες διαμάχης μεταξύ Ταϊβάν και υπηρετικής Κίνας υπάρχει επιτέλους κάποια συνεργασία. Θα έπρεπε να πω ότι οι σχέσεις μεταξύ Ταϊβάν και Ένωσης επίσης είναι θετικότερες τώρα από ό,τι πριν. Η παιδεία και η δημοκρατική διακυβέρνηση στο Ταϊβάν είναι στο επίπεδο της Νοτιού Κορέας και της Ιαπωνίας. Με βάση αυτά τα στοιχεία και άλλα θετικά στοιχεία χαιρετίζουμε την έκθεση του κυρίου Διασδεμέρα και υποστηρίζουμε το αίτημά του για κατάργηση των θεωρήσεων και για τα 27 κράτη-μέλη. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα, οι θεωρήσεις και δεν σημαίνουν ότι δεχόμαστε αλλαγή γενικά του διεθνούς δικαίου ως προς τα εδαφικά δικαιώματα της Κίνας ή του Ταϊβάν. Η Επίτροπος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, η πρόταση για την μεταφορά της Ταϊβάν στο θετικό κατάλογο εγκρίθηκε στις 5 Ιουλίου φέτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια σταθερή αναπτυγμένη δημοκρατία η Ταϊβάν, το ξέρουμε αυτό και πληρούνται όλες οι τεχνικές προϋποθέσεις. Η πρόταση προκύπτει από την περιοδική αναθεώρηση του καταλόγου θεωρήσεων και επί τη βάση των προτάσεων των κρατών μελών ε, αποτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σειρά προϋποθέσεων, αδρομετανάστευση, δημόσια ασφάλεια, mm. αμοιβαιότητα, περιφερειακή συνοχή και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχύσουμε τη συνοχή για την Νοτιοανατολική Ασία και χώρες όπως το Χονγκ το Μακάο, η Ιαπωνία, η ε, Νότιος Κορέα έχουν ήδη απαλλαχθεί από την υποχρέωση θεώρησης ε, και επίσης θέλουμε να βελτιωθούν οι σχέσεις με την υπηρετική Κίνα. Αυτό έχουν αποκατασταθεί απευθεία πτήσεις και υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο για την οικονομική συνεργασία ανάμεσα στην ε, Κίνα και την Ταϊβάν. Και όπως είπατε, η Νότιο Κύπρος, Κορέα, Αυστραλία, η Ιρλανδία ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη χορηγήσει την εξαίρεση και ο Καναδάς ακολουθεί λίγαν συντόμως. Ναι. Ε, φυσικά η εξαίρεση από την υποχρέωση θεώρησης πρέπει να υπακούει στον νόμο της αμοιβαιότητας. Ε, ε, για η, το, Ταϊβάν έχει άρει αυτή την υποχρέωση για μεγάλο κομμάτι των ε, υπηκών πολλών κρατών με της Ευρωπαϊκής Ένωσης. οι Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Κύπροι μπορούν από, τις, από αύριο να ταξιδεύουν ας πούμε χωρίς θεώρηση. Κλείστε τα εισιτήρια σας. Επίση, είναι και θέμα διαμονή ε, που φτάνει μέχρι τι 90 μέρε για του ε, υπηκόου μετά την ε, εξαίρεση από την υποχρέωση θεώρησης. Επίσης, έχουμε τις νήσους ε, Μαριάννη που δεν χρειάζεται να βγουν από τον ανετικό κατάλογο γιατί είναι η Αμερικανική επικράτεια. Είναι εξαιρετικός τρόπος ε, αυτή η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, ούτω ώστε όλοι οι φοιτητές, εργαζόμενοι, ερευνητές να μετακινούνται ελεύθερα και είναι διαδικασία στην απόφαση, το ξέρετε αυτό, Πάντως υπάρχει ευρύτατη υποστήριξη ε, από ό,τι ξέρω στο Συμβούλιο για αυτή την πρόταση. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, μου είπαν ότι στο Κοινοβούλιο υπάρχει εξίσου ευρία υποστήριξη ε, και ε, ευελπιστώ θα υπερψηφιστεί η πρόταση αύριο. Τώρα και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο έχει υποβληθεί πρόταση για την εξαίρεση κάποιων υπηκών της ε, Ταϊβάν γιατί χρειάζονται πρώτερη έγκριση από την Ταϊβάν για να μπουν, εισέλθουν στην Ταϊβάν. Ναι. Οπότε είναι λογικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκλείσει αυτή την ε, κατηγορία των ατόμων που ζουν στο εξωτερικό και είναι κάτοχοι διαβατηρίων βέβαια που έχουν εκτοθεί από τις αρχές ε, της Ταϊβάν. Ε, σας ευχαριστούμε για την συνεργασία, θα έλεγα κλείνοντας ε, και ελπίζουμε ότι με τη νέα συμφωνία θα τονωθούν ήδη πολύ καλές σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσπεταϊβάρ σε πολλούς τομείς όπως το εμπόριο και ο τουρισμός και νομίζω θα είναι υποφιλή συμφωνία για όλα τα μέρη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπο και τώρα ο κύριος Παπα-Νικολάου για δύο λεπτά εξ του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Καταρχά οφείλω να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή και όλου του συναδέλφου που εργάστηκαν για αυτήν την έκθεση. Ε, είναι πράγματι εξαιρετική η εργασία του. Η απελευθέρωση από την υποχρέωση θεώρηση για του κατοίκου Ταϊβάν βεβαίω και είναι προς σωστή κατεύθυνση. Είναι θετικό το γεγονό ότι ξεπεράστηκε το νομικό εμπόδιο που θέτει η μία αναγνώριση της Ταϊβάν από όλα τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, ότι στη βάση της κατά μίαν έννοια αμοιβαιότητας οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα υπόκεινται στο μέλλον στην υποχρέωση θεώρησης κατά την είσοδό τους στην Ταϊβάν, αντίστοιχα δηλαδή με αυτό που κάνουμε και εμείς, για όλες και τις 27 χώρες. Και τρίτον, αποφεύθηκαν οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Στο σημείο αυτό όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου και μία γενικότερη παρατήρηση. Πρόσφατα όλοι γίναμε μάρτυρες τρομοκρατικών ενεργειών όπως η αποστολή παγιδευμένων δεμάτων με εκρηκτικές ύλες από την ελλάδα σε πρεσβείες και σε διάφορες πόλεις της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και από την ιεμένη σε διάφορα κράτη μέλη και βεβαίως όλοι αισθανθήκαμε ότι η ασφάλειά μας απειλείται ποικιλοτρόπως και παντιοτρόπως. Εύλογα, εύλογα λοιπόν όταν οι συμπολίτες μας στην Ευρώπη πληροφορούνται ότι διευκολύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτών τρίτων χωρών, όπως τη Ταϊβάν και άλλες που στο προηγούμενο διάστημα έχουμε εγκρίνει, αναρωτιέται αν αυτό θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο την ασφάλειά του. Στο σημείο αυτό λοιπόν οφείλουμε να απαντήσουμε ότι κάθε φορά που λαμβάνουμε μια τέτοια απόφαση έχουμε προηγουμένως συνεκτιμήσει όλες αυτές τις παραμέτρους γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε τους μηχανισμούς να αντιμετωπίσουμε το όποιο πρόβλημα και να περιφρουρήσουμε την ασφάλεια των συμπολιτών μας και γι' αυτό ακριβώς προχωράμε σε αυτή την απόφαση. Έχουμε συστήματα ανταλλαγή πληροφοριών, έχουμε δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε το όποιο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν καταλήγω και λέγοντας ότι είμαστε ευτυχείς που προχωράμε σε αυτή την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν κάνουμε καμία έκπτωση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των συμπολιτών μας σε όλη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Φαγιόν για δύο λεπτά. Mm. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύρια Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία. Το Ταϊβάν μπορεί να αποτελέσει μια πολύ επιτυχή ιστορία. Μόλις επέστρεψα από εκεί και ε, συνήψα με διάφορες συμφωνίες με την Ένωση και το Ταϊβάν. Γιατί είμαστε ο μεγαλύτερος συνεισφορεύς στην οικονομία τους. Η ανεργία εκεί ανέρχεται μόνο στο 6% και οι σχέσεις συνεχώς βελτιώνονται με την Ένωση, θα αυξηθεί η κινητικότητα, θα έρχονται επισκέψεις τα Ιβανέζων στην Ένωση, ιδίω φοιτητών και φοιτητριών και τα τελευταία χρόνια ιδίως στον οικονομικό τομέα, μερικοί τομείς αντιμετώπισαν δυσκολίες. Αλλά παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι το Ταϊβάν δεν αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες του κόσμου, του αναγνωρίζεται ελεύθερη διακίνηση από 24 από τις χώρες της Ένωσης και επίκειται να καταργηθούν θεωρήσεις και για τις υπόλοιπες μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάστηκε προσπάθεια που την είδαμε και εμείς επί τόπου εκεί ο κόσμος είναι ικανοποιημένος από τη ζωή του και η Ένωση κατήργησε θεωρήσεις και για άλλες χώρες εκτός από το Ταϊβάν και για χώρες των Δυτικών Βαλκανίων εκτός από, τη Βαλκανία και, από την Αλβανία και τη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Έτσι μπορούν και οι χώρες αυτές να γνωρίζουν ότι έχουν ευρωπαϊκή προοπτική γιατί η ελεύθερη διακίνηση είναι από τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ΔΕ Ταϊβάν δεν αντιπροσωπεύει κανένα κίνδυνο για την Ένωση και γι' αυτό κυρίες και κύριοι σας καλώ να ψηφίσετε υπέρ της κατάργησης των θεωρήσεων για το Ταϊβάν για να μπορούν οι πολίτες του να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα η κυρία Βίξτρομ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ έχουμε ένα κατάλογο των τριών χωρών, οι υπήκοοι των οποίων ε, θα πρέπει να έχουν θεώρηση όταν διέρχονται εξωτερικά σύνορα. Υπάρχει ένας άλλος κατάλογος ε, για τους υπήκοους ε, που εξαιρούνται και προσαρμόζονται οι κατάλογοι ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρο. Παραδείγματο χάρη για την Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, έχουμε ήδη ψηφίσει και τώρα σύντομα θέλουμε να καταργήσουμε υποχρέωση θεωρή και για την ε, Ταϊβάν. Η Ταϊβάν έχει ολοκληρώσει μια πλήρη διαδικασία εκδημοκρατισμού, θεσμικές μεταρρυθμίσεις, μια δυναμική κοινωνία των πολιτών ε, και πραγματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτό οδήγησε σε πολιτική σταθερότητα και οικονομική σταθερότητα στην Ταϊβάν. Ε, και ε, υπάρχουν όμως και άλλες αντίστοιχες χώρες στην περιοχή, γιατί νομίζουμε ότι θα υπάρχει μια ομοιόμορφη ζώνη, υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στην ε, περιοχή. Εμείς ε, θεωρούμε ότι ναι, ε, θα ενισχυθούν και οι εμπορικές σχέσεις και οι πολιτιστικές και ερευνητικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ταϊβάν με την κατάργηση της υποχρέωσης θεωρήσεων. Οι υπηκοί της Ταϊβάν δυσκολεύονται ως ιδιώτες να μεταβούν στην Ευρώπη, δηλαδή φοβήθηκαν ε, οι χώρες στην Ευρώπη, όμως δημιουργηθεί ρήξη με την Κίνα. Ε, τώρα βέβαια έχει αλλάξει η κατάσταση ε, και ελπίζω να έχουμε τελειώσει όλα αυτά και να διευκολυνθούν οι πολιτικές επαφές ανάμεσα στους πολιτικούς ηθήνοντες εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, άργουσα τάξη στην Ταϊβάν και ελπίζουμε να ε, βελτιωθεί ο ρόλος της Ταϊβάν γενικότερα στη διεθνή σκηνή. Ε, επίσης, μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ της διαφάνειας και της ενσωμάτωσης όλων, οπότε πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες προς τους γείτονες μας, σε κέρδος, σε συνεργασία και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και πιο ευχάριστο κλίμα σε αυτές τις χώρες. Ε, πάντως, ε, ολόθερμα θα υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση για την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης. Σας ευχαριστούμε. Ο Τσάρλς Τάνοκ τώρα. Κύριε Επίτροπε, εσείς είσαστε πολύ καλοί φίλοι της Ταϊουάν από την εποχή που ήσασταν ε, ευρωβουλευτής. Και εγώ είμαι πρόεδρος της ομάδας φιλίας με την Ταϊουάν και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ενθουσιάζομαι με την ευκαιρία αυτή που θα μπορούν να έρχονται οι Ταϊβανοί αλλά και οι Ταϊβανέζες στη ζώνη του Σέγγεν χωρίς να χρειάζονται βίζα. Αυτό το λέτε εσεί φιλελευθερωποίηση προψαϊκή θεώρηση. Η χώρα μου και η Ιρλανδία, που είναι βέβαια εκτό Σέγγεν, έχουν ήδη δώσει στου ε, πολίτε στη Ταϊβάνη τη δυνατότητα στη Ταϊβάνη το δικαίωμα να έρχονται χωρί βίζα εδώ και 1,5 χρόνο ήδη. Και το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του επιχειρηματικού τουρισμού έχει δικαιολογήσει αυτή την απόφαση που ήταν πολύ θετική. Η Ταϊβάν είναι μια ανθούσα και ε, πολύ σημαντική δημοκρατία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημιουργεί ειρήνη και ευμάρεια στην περιοχή της. Μπορούμε όλοι να ευνοηθούμε από το να έχουμε καλύτερες εμπορικές σχέσεις με την Ταϊβάν και την οικονομία της η οποία ενισχύεται κάθε χρόνο με μεγάλη οικονομική μεγέθυνση και είναι ένα εφαλτήριο για επενδύσεις στην Κίνα. Η Ευρώπη βέβαια σιγά σιγά γίνεται έρχεται στο ίδιο επίπεδο σαν τόπος προορισμού για τους φοιτητές και τους ερευνητές από την Ταϊβάν. Και είναι λοιπόν θετικές αυτές οι επαφές με κάθε τρόπο. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την ε, αλληλεγγύη μας και την υποστήριξή μας με τη Ταϊβάν, η οποία με την φωτισμένη ηγεσία που έχει, έχει καταφέρει να βγει από τον αποκλεισμό στον οποίο τον είχε βάλει η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. 1,5 λεπτό κύριος Βοργέζιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος πολύ καλά έχει χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του και τις ικανότητές του να δώσει μια, για να δώσει μια αυστηρή αλλά δίκαια ε, πρόταση. Να μπορέσουν λοιπόν να εξασφαλίσουν, να εξασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών της Ταϊβάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Εγώ δεν είμαι σίγουρος για αυτό που έχει γίνει για χώρες όπως η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη και η Αλβανία για τις οποίες ήρθε η ανάγκη βίζας και ορισμένοι μιλάνε και για την Τουρκία σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ λοιπόν επικροτώ την ε, πρόταση του κ. Σουέγρα και την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι φανερό ότι θα είναι θετική. Όλοι, θεωρούμε, τι, όλοι γνωρίζουμε τι ήταν η Κίνα για πάρα πολλές δεκαετίες όταν ήταν η, είχε το όνομα Εθνικιστική Κίνα. Ήταν υπέρμαχος της και αντιμετώπισε μεγάλες απειλέ Υπήρξαν τότε και προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά Γνωρίζουμε ότι τώρα οι Κίνες της Ταϊβάν είναι καλόδεκτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στις σχέσεις με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σαφές ότι υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα ενσωμάτωσης των πολιτών της Ταϊβάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα με άλλες χώρες, η Ταϊβάν δεν θίγει τα δικαιώματα της, ε, των μειονοτήτων, θρησκευτικών και εθνοτικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλόδεκτοι λοιπόν στην ε, Ταϊβάν και ιδίως οι πολίτες της Παδανίας. Ο κ. Κόβατς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως ε, το σύστημα των θεωρήσεων είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να αποφευθεί η λάθρο μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η λαθρεία διαμονή στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν εξετάζουμε αυτό το θέμα του θετικού και του αρνητικού καταλόγου, οφείλουμε να εξετάζουμε κατά περίπτωση τι συμβαίνει η δημόσια τάξη, στην εν χώρα, η εξωτερικές τις σχέσεις, η αμοιβαιότητα, αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να λειτουργεί καλά και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις χώρες. Αλλά δεν μπορεί κάποια χώρα να μπει στον θετικό κατάλογο παρά μόνο αν πληρούνται όλα τα κριτήρια. Τρεις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται ακόμη θεώρηση ε, για ε, την Ταϊβάν. Και περιμένουμε τα, ε, τις προτάσεις ε, των κρατών μελών δυστυχώς για να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα προβλέπεται από τη διαδικασία, δεν είναι χριστουγεννιάτικο δώρο προς την ε, Ταϊβάν η κατάργηση της θεώρησης. Η κυρία Γκέντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάργηση των θεωρήσεων για τους πολίτες του Ταϊβάν είναι κάτι που το χρωστούσαμε στη χώρα αυτή από πολύ καιρό. Είναι σημαντικός εμπορικός μας εταίρος. Και άλλοι το ίδιο σημαντικοί εταίροι έχουν ήδη πάρει το δικαίωμα αυτό. Το Ταϊβάν είναι λοιπόν πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος, ο τέταρτος στην Ασία εταίρος μας και αναμένουμε οι εμπορικές αυτές σχέσεις να αναπτυχθούν περαιτέρω. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα, στην ανάπτυξη και επομένως η κατάργηση των θεωρήσεων είναι κάτι που μπορεί να συμβάλλει ακόμη περαιτέρω στην ανάπτυξη στους τομείς αυτούς των σχέσεων. Αναμένουμε από τους εταίρους μας να καταργήσουν και εκείνοι τις θεωρήσεις για όλες τις χώρες της Ένωσης και οι τρεις χώρες τις που ακόμη επιβάλλουν θεωρήσεις για τους πολίτες της Ταϊβάν πρόκειται σε λίγο να τις καταργήσουν και εκείνες. Το Ταϊβάν έχει γίνει πολύ πλούσια χώρα ενώ οι απαρχές της ήταν πολύ πτωχές και επειδή δεν υπάρχουν και μεταναστευτικές ροές δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε από το Ταϊβάν. Δεν βλέπω ούτε τον κύριο Ομπερμάγερ, ούτε την κυρία φλάση Κοβαμπένοβα Δεν είναι παρόντες. Γι' αυτό περνάμε στην οφθαλμοθυρία. Και βλέπω εδώ την κυρία Άντλικεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Υποστηρίζω απόλυτα αυτά που είπαν οι εισηγητέ Δία Δεμέρα και η κυρία Κόβατσεφ. Το Ταϊβάν είναι ανεπτυγμένη χώρα και προφανώς πληρεί τα ανώτατα κριτήρια ασφαλείας και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω προς τους συναδέλφους ότι θα έπρεπε να εγκρίνουν την κατάργηση των θεωρήσεων για τους πολίτες της. Είναι επίσης μέλος του ΠΟΕ. Δεν πρέπει όμως να σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να ζητήσουμε την ένταξη του Ταϊβάν και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας ή την Διεθνή Οργάνωση για τις Κλιματολογικές Αλλαγές. Είναι χώρα που αξίζει τέτοια αναγνώριση γιατί είναι σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Ασία. Η ανάπτυξη τέτοιων σχέσεων θα ωφελήσει και τα δύο μέρη. Και αναμένουμε ανάπτυξη περαιτέρω των σχέσεων. Οι διαπραγματεύσεις για ένα πιο ολοκληρωμένο εμπορικό πλαίσιο συνεργασίας με το Ταϊουάν θα ήταν επίσης κάτι το θετικό. Αν κινηθούμε προς εκείνη την κατεύθυνση, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι η κατάργηση των θεωρήσεων είναι σημαντικό βήμα. Ευχαριστώ. Κύριος Ζεντσιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι. Θέλω καταρχά να συγχαρώ τον συνάδελφό μας Δίας Μέρα για την έκθεσή του. Είμαι βέβαιος ότι θα εγκριθεί ομόφωνα, ομόφωνα. Θα ήθελα να αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν στηρίζει την αρχή της αμοιβαιότητας στις σχέσεις της με τρίτες χώρες. Το Ταϊουάν θα τύχει εξαίρεση από την υποχρέωση των θεωρήσεων εκ μέρους όλων των χωρών της Ένωσης και με τη σειρά του θα καταργήσει τις θεωρήσεις για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κύπρο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όμως δεν κάνουν κάτι ανάλογο για τη Ρουμανία. Και μάλιστα θα έλεγα, ε, πρέπει να πω, ότι επέβαλαν και αύξηση της τιμής των θεωρήσεών τους. Η Ένωση εδώ πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο με πλήρη αμοιβαιότητα Όσο είναι αρμοδιότητά της η θεωρήσεις, πρέπει να παίρνει μέτρα για να λύνει τέτοια προβλήματα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μιγκάλσκι. Ευχαριστώ. Επίτροπο, όπως βλέπετε, υπάρχει συνένεση στην αίθουσα. Μπορεί να μην εγκριθεί με ομοφωνία η έκθεση, αλλά σίγουρα θα υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία. Μεγάλη υποστήριξη από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα σχόλια που ήδη ακούσαμε. Προφανώ η Ταϊβάν κληρεί όλα τα ε, κριτήρια οικονομικά και πολιτικά ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να ε, ισχύσει η εξαίρεση από την υποχρέωση θεώρησης. Μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα, δηλαδή ο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δημοκρατικής κοινωνίας, ε, πορείας προς εκδημοκρατισμό που ολοκλήρωσε η Ταϊβάν. Πέρα από την οικονομική επιχειρηματολογία, όπως ε, σωστά είπε ο κύριος Μπορκέτσιο, δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε την πολιτική διάσταση. Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι θέμα και γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε τους, ε, ε, την Ταϊβάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ταϊβάν έρχεται στο θετικό κατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτε τη Ταϊβάν μπορούν να έρχονται χωρί υποχρέωση βίζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτού του ανθρώπου. Αλλά η πολιτική είναι δούνε και λαβίν. Αλή βερίσ και θα ήθελα αυτό να σημαίνει και αμοιβαιότητα για του πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν και αυτοί να πηγαίνουν στην Ταϊβάν. Μέχρι στιγμή αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η Ταϊβάν είχε απλώ δηλώσει την ε, πρόθεσή τη μέχρι το τέλο του χρόνου να γίνει αυτό πραγματικότητα. Ελπίζω ότι αυτή η πραγματικότητα, αυτή η πρόθεση, συγγνώμη, μάλλον θα υλοποιηθεί. Και θα υποστηρίξω λοιπόν εάν την πρόταση του εισηγητή αν πράγματι η Ταϊβάν όπως είπε ο εισηγητή, από αύριο έχει εξασφαλίσει την είσοδο των πολιτών τη Ευρωπαϊκής Ένωση χωρίς βίζα στο εδαφό. σα. ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρος. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επίτροπο Μέλστρομ να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή και όλους εσάς για την ευρεία υποστήριξή σας, για την πρόταση μεταφοράς της Ταϊβάν στο θετικό κατάλογο. Ε, θα ήθελα να καθυσυχάσω τους συναδέλφους που έχουν ακόμη κάποια ερωτηματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ μεθοδικά ε, εξετάζει κάθε μεμονωμένη περίπτωση. πρωτού υποβάλει τέτοια πρόταση εξαίρεση σας διαβεβαιώ ότι ήμασταν πάρα πολύ σχολαστικοί. Επίσης, προς τον τελευταίο μιλτή θα ήθελα να πω ότι αύριο θα γίνει αυτό και για τις υπόλοιπες χώρες. Από αύριο θα αρχίσει να ισχύει αυτό. Υπάρχει αμοιβαιότητα. Μετά την αυριανή ψηφοφορία θα στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα μπορούμε να ελπίζουμε σε ακόμη καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στο λαό της Ταϊβάν και τους λαούς της Ευρωπαϊκής Να Σας ευχαριστώ όλους για μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, ο κύριος Δίας Δεμέρο, εισηγητής μας. Μερσή κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Δίας Δεμέρο. Η ευγένεια υποχρεώνει. Γι' αυτό πρέπει εγώ να εκφράσω την απεριόριστη μου εκτίμηση σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι από τις διάφορες πολιτικές ομάδες έχουν υποστηρίξει την ε, έκθεσή μου. Την έκθεση που είχα την τιμή να παρουσιάσει τα ποινότητά μου. Επίση ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι βοήθησαν την εργασία μου. Δεν θα ήταν δίκαιο όμω να παραλείψω να πω ότι ο, ο κύριος υπεύθυνο για όλα αυτά ή κύρια υπεύθυνο είναι η ίδια η Επίτροπος Μέλστρομ η οποία με την υποστήριξή τη, με τον ενθουσιασμό τη και με την θαυμάσια ε, ομάδα της έκανα δυνατό να προωθηθεί αυτό το θέμα και αυτό ήταν φυσικά και μια πράξη αποδόσης δικαιοσύνης για μένα. Όταν πέραν αυτών που είπα λοιπόν κύριε Πρόεδρε θέλω να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου και προς το λαό της Ταϊβάν, τις αρχές της Ταϊβάν και φυσικά στη θαυμάσια ομάδα διπλωματών και διπλωματριών που έχει περηφάνη σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδίω στι Βρυξέλλε. Τίποτα άλλο και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δία Στεμέρα. Έχει κλείσει η συζήτηση λοιπόν και θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή αύριο αν θέλει ο Θεός βέβαια.